Ναι, συνάδελφοι. Σας ε, καλωσορίζω όσους ήρθαν στην ώρα τους, οι οποίοι βεβαίως δεν πρέπει να τιμωρηθούν και όλα που ήρθαν στην ώρα τους, οπότε ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά. Ο Παλ Ρούμπιχ είναι ο εισηγητής και θα τον παρακαλούσα να ξεκινήσει και μπορούν μετά οι συνάδελφοι να πάρουν τον λόγο. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρόιλ, κυρίες και κύριοι. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι ένας δυσνόητος τομέας για πολλούς, αλλά από την άλλη είναι η ιδιοκτησία κάτι το πολύ σημαντικό σε μια οικονομία και όπως ακριβώς η φυσική ιδιοκτησία είναι σημαντική, το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική ιδιοκτησία και η προστασία της πνευματικής ε, ιδιοκτησίας ε, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και ακόμα και στις χώρες του πρώην ε, κομμουνισμού όπου δεν ήταν πολύ ψηλή προτεραιότητα. Να γνωρίζετε τώρα πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν οι ιδέες και η καινοτομία και να υπάρξει έτσι επιτυχία στην οικονομία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολο από 27 κράτη-μέλη να δημιουργηθεί ένας ενιαίος οικονομικός χώρος, ένας οικονομικός χώρος ο οποίος πρέπει να είναι χωρίς σύνορα, ελεύθερος από τα πολιτικά και γεωγραφικά σύνορα και η έννοια βεβαίως της εσωτερικής αγοράς έχει ιδιαίτερη σημασία και για την πνευματική ιδιοκτησία και βεβαίως οι άδειες ε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι άδειες αυτές ε, έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία ειδικά όσον αφορά το copyright σε πολλούς ε, τομείς παίζει ένα σημαντικό ρόλο ανεξαρτήτως του πώς ε, δίνονται οι άδειε. Αυτό το πώς δίνονται δηλαδή οι άδειε είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην Ευρώπη και παγκοσμίω και εδώ πέρα νομίζω απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τις ε, δομές της, ε, να τις εντείνει και όσον αφορά επίσης και την εφαρμογή. Το θέμα εδώ δεν είναι μόνο οι μεγάλες διεθνείς εταιρείε που πρέπει να προστατεύσουν ε, εξελίξεις ε, πολλών ε, ετών γιατί μετά αντιγραφής οι δεν έχουν αυτό το κόστος της έρευνας και της καινοτομίας αλλά ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις ή τις μικρές επιχειρήσεις είναι πάρα... και για τους εφευρέτες είναι πάρα πολύ σημαντικό να απολαμβάνουν την προστασία των δικαστηρίων και να προστατεύεται η ιδιοκτησία τους. Γι' αυτό, αυτό το οποίο λέω πρώτο είναι πως θα πρέπει να δούμε την διαθεσιμότητα η οποία θα πρέπει να προωθηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η πνευματική ιδιοκτησία θα πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την εσωτερική αγορά και το ίδιο και η άδεια. Αυτό βεβαίως ισχύει και πρέπει να το σκεφτούμε ιδιαίτερα στο πλαίσιο των γλωσσών και να δούμε τι γίνεται με τις άδειε πέραν των γεωγραφικών συνόρων όσον αφορά τις γλώσσες, δηλαδή να δίνονται άδειε για τα γαλλικά, για τα ισπανικά, για τα γερμανικά, έτσι ώστε να ισχύουν διασυνοριακά και με ένα γλωσσικό μοντέλο και όχι μόνο εντός της Ευρώπης αλλά παγκοσμίως. και να σκεφτούμε έτσι παγκοσμίω αν θα μπορούσαν να ισχύσουν για ένα παγκόσμιο γλωσσικό καθεστώς αυτές οι άδειε. Και εντό Ευρώπη βεβαίω αυτό θα ενίσχυε πάρα πολύ τα, τα πράγματα και τι εγγυήσει που δίνονται. Το τρίτο σημείο αφορά την διαλειτουργικότητα και την τεχνολογική ουδετερότητα και αυτό θα συνεισφέρει στο ότι το περιεχόμενο θα μπορεί μετά να διανέμεται σε πάρα πολλές πλατφόρμες και μορφές και να υπάρχει όπως είπα αυτή η τεχνική ουδετερότητα. Ειδικά αυτό ισχύει στην πληροφορική και στις ε, τεχνολογίες των πληροφοριών. Εδώ πέρα ακριβώς θα πρέπει να δώσουμε βάρος. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το σημείο 4, σημαντικό θα ήταν να υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα απευθύνονται, ειδικά αν μιλάμε για πανευρωπαϊκές ε, άδειε να υπάρχει μία υπηρεσία η οποία θα γνωρίζει την κατάσταση και στα 27 κράτη-μέλη και πιθανώς θα είναι στην διάθεσή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων, επιβολή των δικαιωμάτων και εκτός της Ένωσης για ευρωπαϊκές όμως γλώσσες, δηλαδή να προσπαθεί τις ευρωπαϊκές γλώσσες ε, να τις επιβάλλει και να τις προστατεύει και εκτός της Ένωσης. Σημείο θα έπρεπε να μελετήσουμε κύρωσης ε, για παραβιάσεις όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού, όχι μόνο για τις ζημιές, αλλά και για την αποκατάσταση και για τις απώλειες που σημαίνουν αυτές οι ζημίες και η πρόληψη νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ πέρα και το σημείο 6 είναι το σημείο των κυρώσεων βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και εμπορίου που γνωρίζουμε ούτως ή άλλως πως ε, το δίκαιο του ανταγωνισμού μπορεί να επιφέρει πάρα πολύ υψηλε ποινές ε, και είναι βεβαίως ζήτημα το οποίο ανοίξει την εκτελεστική αρμοδιότητα της Κομισιόν και στο, νομίζω στο μέλλον θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μοντέλο αυστηρότερης παρέμβασης ειδικά σε αγορά και πειρατεία προϊόντων για να είναι η αντίδραση γρήγορη και αποτελεσματική μαζί με τις ελληνιακές αρχές. Για την ε, Κομισιόν και για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σημαντικό είναι να γίνεται πάντα αξιολόγηση αντικτύπου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί βεβαίως αν μιλάμε για μια μεγάλη επιχείρηση έχει πολλές περισσότερες δυνατότητες ε, και προσφυγής και αντίδρασης, αλλά είναι πολύ προβληματική κατάσταση για μια μικρή επιχείρηση. Οπότε πρέπει να δούμε την αξιολόγηση του αντικτύπου όπως προβλέπεται και στο σχετικό νομοθέτημα και πρέπει αυτό να γίνει κατά προτεραιότητα. Τέλος, με την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου, Παρατηρητηρίου για την Παραποίηση και την ε, Πειρατεία θα πρέπει να αναπτυχθούν προτάσεις ε, για κοινά κριτήρια και τυποποιημένες ε, διαδικασίες για συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά για το τι μπορεί να γίνει για την παραποίηση και την πειρατεία και βεβαίω πρέπει να υπάρχει και μια διαφάνεια για να υπάρχει και αυτή η αποτροπή, αυτός ο αποτρεπτικός χαρακτήρας. Και έτσι βεβαίως θα έχουμε τις θετικές οικονομικές εξελίξεις που θέλουμε στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Από πλευρά των σκιωδών εισηγητών θέλει κάποιος τον λόγο. Ρίβαζη, λοιπόν, έχει τον λόγο. Frau correct? Λάθος το λέω. Ναι, εσείς, εσείς έχει τον λόγο. Ε, έχω λάθος όνομα εδώ, συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Ε, εν πάση έχει το λόγο. Και με Νόμιζα ότι είπατε να μιλήσουν πρώτα οι σκιώδεις ηγητές. Δεν είμαι σκιώδης ηγητρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρουμπίχ για την πρόταση έκθεσή του. Πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω καλύπτει όλα τα σημεία που ενδιαφέρουν την Επιτροπή Βιομηχανίας. Μόνο στο σημείο 6, και που λέει να κάνει πλήρη χρήση των κυρώσεων που έχει στη διάθεσή της ε, σε σχέση με το δίκαιο περί ανταγωνισμού και εμπορίου, γιατί να μην προσθέσουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα ενημέρωσης για παράδειγμα. Γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ ε, ευαίσθητο, πολύ λεπτό και δυσεπίλητο. Καμία κυβέρνηση δεν έχει βρει μια λύση αυτή τη στιγμή να διασφαλίσει δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων copyright, πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων δημιουργού και των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, των χρηστών και κυρίως το θεμελιώδες και αναπαρατήρητο δικαίωμα της ενημέρωσης. Κατά του λοιπού συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητού Ρουμπίχ. Ευχαριστώ. Herzlichen Dank, Frau Kutsche. Gibt es weitere Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη, γιατί θεωρώ πως η έκθεση Ρούμπιχ πηγαίνει σε μια εξαιρετική κατεύθυνση και τα σημεία τα οποία οπωσδήποτε θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια νομίζω αναφέρονται εδώ και πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις ε, ποιες θα είναι αυτές οι ποινές κτλ. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε κάποιες ε, προτάσεις ε, και μετά βεβαίως θα τα δούμε όπως είπαμε σε επιτροπές και καθ' όλη τη διάρκεια της ηττίας. Σε πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ με αυτή τη γνωμοδότηση με την οποία συμφωνώ πλήρως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Καλημέρα. Οι πράσινοι έχουν να θέσουν δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην ίδια ομάδα την παραβίαση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας που μπορεί να αφορά το, την υγεία από τη χρήση που κάνει κάποιος που μπαίνει στο ίντερνετ και κατεβάζει παράνομα μια ταινία ή, μια, ή ένα τραγούδι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεύτερον, να επανεξετάσουμε το θέμα των διπλωμάτων εν γέννη το κόστος τους, το κόστος κατοχύρωσης τους δηλαδή, διότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει καταχρηστική χρήση των ε, ε, διπλωμάτων αυτών ή δικαστική εκμετάλλευση, δικαστική παρέμβαση για την εκμετάλλευση αυτών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθιστώντας πολύ δύσκολο να μπουν κάποιοι άνθρωποι στην αγορά των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μπορεί να υπάρχουν βεβαίως και καταχρήσεις. Σας ευχαριστώ να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο Στανκίκας. Yes. Thank you very much for, for your opinion, for your Ευχαριστώ για την γνωμοδότησή σας για αυτό το θέμα το πολύ ευαίσθητο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των παραποίησης, πειρατείας κτλ. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσάρμοσε την ανακοίνωσή τη σε θέματα εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία και ε, θεσπίσαμε πολλά μη νομοθετικά μέτρα που συμπληρώνουν τα νομοθετικά μέτρα που ήδη διαθέτουμε. Για παράδειγμα, η, η οδηγία περί εφαρμογή, ε, ο κανονισμό, ο σχετικό και αυτά τα μη νομοθετικά μέτρα, επαναλαμβάνω, συμπληρώνουν τα προηγούμενα νομοθετικά μέτρα. Το πιο σημαντικό είναι η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Απομίμηση και την Πειρατεία. Και επισημάναμε τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των σωματείων τους, γιατί συμμετέχουν στο νέο αυτό παρατηρητήριο. Το παρατηρητήριο άρχισε με τη μελέτη των εφισταμένων δεδομένων και επεξεργάζεται στοιχεία και τις γνώσεις που συγκεντρώνουμε για θέματα απομίμησης και πειρατείας. Κατόπιν ε, θα καταρτίζει τη ΣΥΟΣ έκθεση, το παρατηρητήριο, προκειμένου να μας βοηθάει στη λήψη αποφάσεων πολιτικής. Επίσης θα προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών το παρατηρητήριο αυτό, αλλά και μεταξύ των διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας και μεταξύ των εταιριών. Σας ευχαριστώ πολύ για την γνωμοδότηση. Ε, ευχαριστώ. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Να σας υπενθυμίσω προθεσμία 25 Φεβρουαρίου για τροπολογίες και 17 Μαρτίου, εάν όλα πάνε καλά, θα ψηφίσουμε. Περνάμε στο σημείο 6. Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συνεργειών ε, για την έρευνα και την καινοτομία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 7 Πρόγραμμα Πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη κτλ. λοιπά Ένα ε, μακροσκελής τίτλος εδώ πέρα τον διάβασα γιατί ο κύριο συνάδελφο εδώ πέρα δεν έχει έρθει ακόμα στην αίθουσα ο εισηγητή. Οπότε έλεγαν πω ε, έρθει ο κύριο Χατζημαρκάκης. Ελπίζω από στιγμή σε στιγμή να έρθει. Δεν ξέρω ε, αν έχει νόημα να μιλήσει κάποιο άλλο πριν τον εισηγητή. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι, δύο λεπτά. Μη φύγετε όμω. Μη φύγετε. Συνεχίζουμε σε λίγο. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht weiter. Mit besonderer Freude begrüßen wir den Kollegen Chachi Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζουμε με χαρά τον κύριο Χατζη Μαρκάκη, σημείο 6. Δεν το ξαναδιαβάζω, γιατί τα έχουμε πει όλα. Είναι λοιπόν η έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συνεργειών Όταν ε, είναι έτοιμος λοιπόν και έχει αναλάβει τις δυνάμεις του μπορεί να ξεκινήσει να μας πει τα σχετικά. Ε, με συγχωρείτε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και εσείς είστε κατά του κλονισμού οπότε δεν μπορώ να στείλω εδώ πέρα τον, τον κλόνο μου για να ξεκινήσει η θέση μου. Εν πάση περιπτώσει να αναφερθώ εδώ πέρα στην αλλαγή των ε, παραδειγμάτων, των, των ε, μοτίβων, γιατί αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα για την ε, περιφερειακή πολιτική αφενός που δεν μας αφορά βέβαιως αλλά για την ε, καινοτομία που όντως μας αφορά είναι μια αλλαγή θα έλεγα των κυρίαρχων παραδειγμάτων που έχει ήδη εν μέρος ε, λάβει χώρα. Ήδη στα παλαιά ερευνητικά προγράμματα γύρω στο 25% του ποσού που πήγαινε στα περιφερειακά ταμεία αφιερώνονταν στην έρευνα στην ε, καινοτομία και εκεί πέρα όπου γίνονταν αυτό πραγματικά είχε καρποφορήσει και είχε σημαντικές επιτυχίες και αυτό βεβαίως ε, και ε, οδήγησε και εμένα και τον κύριο Φανίστελ Ρόι να θεωρήσουμε πως πρέπει να πάμε ακόμη εντονότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Το ακούμε παντού πως αυτό το κοινοβούλιο υποστηρίζει όλα τα μέτρα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της κλιματικής αλλαγής. Αλλά εάν το κάνουμε αυτό, εάν ε, θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια κλιματική πολιτική, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διάθεσή της ε, και αυτά τα οποία μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικότερα είναι αυτά τα οποία έχουν την περισσότερη χρηματοδότηση, δηλαδή Ταμείο Συνοχής ε, και πρόγραμμα πλαισίου και αυτά τα οποία πηγαίνουν και στην ε, γεωργική πολιτική και στην ανάπτυξη της υπαίθρου γιατί φεύγουμε απευθείας από την άμεση ενίσχυση των αγροτών στην ενίσχυση γενικά της υπαίθρου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτά εδώ πέρα. Πριν πρόκειται λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε διαφορετικά μέσα ενίσχυσης όπως παραδείγματο χάρη το ΣΥΠ, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία ή το πρόγραμμα πλαίσιο 7 το μεγαλύτερο του κόσμου, το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα του κόσμου με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές οδηγίες Δηλαδή ο κάθε ένας ο οποίος κάνει αίτηση πρέπει να συμπληρώσει πάρα πολλά διαφορετικά έντυπα και δεν υπάρχει κάποια συμμόρφωση με αυτά τα οποία γίνεται στην περιφερειακή και διαρθρωτική πολιτική και τα κράτη-μέλη εκείνα στην Ευρώπη τα οποία είναι ιδιαίτερα εφευρετικά μπορούν να οδηγηθούν σε τέτοιες συνέργειες αυτά τα οποία όμως δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και τι λέμε εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πιο ενιαία κριτήρια ενίσχυσης της ερευνητική πολιτικής Αφενό και της περιφερειακή πολιτική αφετέρου. Είναι απλούστερο δηλαδή να έχουμε συνέργειες, αλλά ταυτόχρονα και στην διαμόρφωση των στόχων της πολιτικής να ενισχύσουμε ιδιαίτερα στον τομέα έρευνα και καινοτομία. Ξέρετε πως ε, ως Ευρωπαίοι θα είμαστε παγκοσμίως αγωνιστικοί αν πάμε μόνο προς αυτή την ε, κατεύθυνση και αναλόγως πρέπει να κατευθύνουμε και τα μέσα μας. Και μόνο έτσι εξηγείται το ότι κάποια κράτη-μέλη πράγματι έχουν αναπτύξει κάποια κλάστερ, κάποιους πόλους αριστείας, είτε μιλάμε για την ανοτεχνολογία στο Ζάρλαντ, παραδείγματο χάρη στην πατρίδα μου, όπου θεωρείται ότι είναι η περιοχή η οποία είναι πρώτη στην στην ανοτεχνολογία, είτε μιλάμε για την πληροφορική και ήταν περιοχές οι οποίες παλαιότερα είχαν μείνει πίσω και κατάφεραν να βρεθούν στην κορφή με την χρήση ακριβώς αυτών των μέσων. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα μας Πρέπει λοιπόν να γίνει έτσι μια απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Απλά να υπενθυμίσω κάτι το οποίο δεν ήταν ε, στο προσκήνιο του προγράμματος πλαισίου 7 και θα πρέπει να έρθει στο πλαίσιο πρόγραμμα 8. Πρέπει να ενισχύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν και καλή διαχείριση γιατί συνεχώς μιλάμε για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτό γίνεται μόνο σε ένα βαθμό. Εκεί πέρα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να τα διοικηθούν αυτά. Τώρα δεν θέλω να κάνω μαθήματα εδώ πέρα, αλλά πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινητοποιηθεί τα άτομα αυτά τα οποία βρίσκονται στις περιφέρειες και λαμβάνουν ή ζητάνε τέτοια χρήματα θα πρέπει να ε, κάνουν κάποια εκπαίδευση, να έχουν κάποια εκπαίδευση για να είναι πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την χρήση αυτών των μέσων. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε από τα κλάστερ να οδηγηθούμε σε ένα ενιαίο τοπίο έρευνας και στην Ευρώπη και τα μεγάλα θέματα τα οποία συζητάμε στην Επιτροπή μας, ε, αποτελεσματικότητα και στις συγκοινωνίες αυτό γίνεται με τις υποδομές αφενός, αλλά και με την έρευνα και την καινοτομία, με το να συγκεραστούν αυτά τα στοιχεία. Με το να έχουμε βεβαίω υποδομές, ευρυζωνικότητα, έχουμε κάνει μια συζήτηση και θα την κάνουμε και αυτή τη βδομάδα για τις επικοινωνίε και βλέπουμε πως οι φιλοδοξίες μας δεν κάνουν τίποτα πύχη στην ηλεκτρική κινητικότητα εάν δεν υπάρχει παραδείγματο χάρη η απαραίτητη υποδομή. Η υποδομή σημαίνει λεφτά σε νέε ιδέες. Και αυτή είναι η προσέγγιση μου και ευχαριστώ και τον κύριο Φανίστελ Ρόι ο οποίος είναι και εδώ πέρα και στην Επιτροπή Περιφερειακών ε, Θεμάτων από το ΕΛΚΑ και θέλω να τον ευχαριστήσω και για την ε, πρωτοβουλία και για το πόσο παρακολουθεί αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Θέλει κάποιον λόγο. Βίνκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την έκθεση του κυρίου Χατζημαρκάκη και τον ευχαριστώ πράγματι και εγώ μπορώ να υπογραμμίσω πως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις περιφέρειες και για εμάς ε, το κομμάτι της ε, συνοχής ε, και της περιφερειακής ενίσχυσης ε, το οποίο πηγαίνει στην έρευνα πρέπει να αυξηθεί. Πράγματι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα πως δεν λειτουργεί σωστά η απορρόφηση ή η ροή. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να συντονιστούμε και καλύτερα. Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι ε, εμπλέκονται και εργάζονται με τελείω διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές αλλά παράλληλα ο ένας τον άλλον χωρίς να συναντιόνται και δεν συνεννοούνται και δεν γνωρίζουν τι θα μπορούσε να συνδυαστεί και είναι άρα πάρα πολύ σημαντικό πως χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που διοικούν όπως είπατε τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας αλλά πράγματι πρέπει να έχουμε ενιαία κριτήρια για την διοίκηση, την διαχείριση αυτών των ε, προγραμμάτων έρευνας και γενοτομίας και πράγματι πρέπει να γίνει αυτή η έκκληση για να διασφαλίσουμε πώς θα υπάρξει μια απλοποίηση και να υπάρξει μεγαλύτερη ροή αυτών των κονδυλίων στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Χαίρομαι επίσης για το ότι ζητάτε εδώ πέρα και παρατηρείτε μια μεγαλύτερη ροή μέσω των διαρθρωτικών ε, ταμείων και συμφωνούμε με αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η βασική κατεύθυνση αυτής της γνωμοδότησης με βρίσκει σύμφωνο. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω μόνο. Πρώτα απ' όλα, σημείο 1. Δεν είμαι σίγουρος όσο και αν αγαπάμε την πατρίδα μας και τις περιφέρειες και την τοπική οικονομία και την έρευνα, δεν είμαι σίγουρος εάν σε κάθε περίπτωση γίνεται αποτελεσματικότερα σε περιφερειακό επίπεδο η καινοτομία. Κάποιες ε, καινοτομίες χρειάζονται λίγο μεγαλύτερο πλαίσιο. Δεν ξέρω. Εδώ θα έπρεπε να είναι κάπως πιο ευέλικτη η διατύπωση. Δεύτερον, καλό θα ήταν και εδώ ο συνάδελφος ε, το ανέφερε εάν αυτή η καινοτομία θα έπρεπε εδώ να αναφερθεί, δηλαδή να αναφέρουμε μια αηφόρο οικονομία ως πρότυπο και νομίζω καλό θα ήταν να κατονομάσουμε αυτές τις καινοτομίες που είναι σημαντικές για την νέα αυτή βιομηχανική επανάσταση θα μπορούσαμε να το συμπληρώσουμε. Κατά τα λοιπά, νομίζω είναι πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας πω ότι καταρχάς υποστηρίζω πλήρως ε, την εξαιρετική έκθεση του κύριου Χατζημαρκάκη. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Χρειαζόμαστε μια καλή έκθεση, ένα καλό κείμενο επίσης από την Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιατί αν δούμε την κατάσταση θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Το πού θα βρούμε νέα κονδύλια για την κοινοτομία δεν εμφανίζεται, δεν υπάρχει σε πολλές περιφέρειες. Οι δυνατότητες να υποβληθούν αιτήσει είναι περιορισμένες σε πολλές περιοχές. Βέβαια, αυτό υπάρχει και πρόβλημα ενημέρωση από πλευρά των ταμείων. Η ρευστότητα τη χρηματοδότηση αποτελεί τεράστιο πρόβλημα. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι μικρέ επιχειρήσει γενικά, τα μικρά πανεπιστήμια δεν μπορούν εύκολα να μετέχουν σε, τέτοιες, ε, σε τέτοιου αγωνισμού διότι υπάρχει συγχρηματοδότηση. Αυτό δεν είναι κακή ιδέα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ρευστότητα που είναι ευθεία, ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία καθυστερεί και πληρώνει στο τέλος πάντα. Ζητά πάντα από τους μικρότερους εταίρους να καταβάλουν πρώτοι τα κονδύλια. Αυτό είναι ένας άλλος προβληματικός τομέας. Υπάρχουν επίσης κράτη-μέλη που δεν καταβάλουν πλήρως το τμήμα της χρηματοδότησης που τους ανήκει. Δεν ξέρω πώς ε, λειτουργούν τα νούμερα. Βάζεις ένα ευρώ και παίρνει δύο. Ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και με τα κράτη-μέλη γραφειοκρατία. Είχαμε μια μήνυα κρόαση για το θέμα αυτό. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύω ότι η ιδέα του να υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια άτομα που γίνονται ειδικοί ακριβώς για αυτή τη διαδικασία δεν είναι κακή. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι καλή χρήση κονδυλίων και χρόνου να μαθαίνουν όλοι όλες τις λεπτομέρειες των αιτήσεων. Να λοιπόν ένα τομέα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε προσεκτικότερα. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τις περιφέρειες να έχουν μια στρατηγική για τον τομέα αυτό. Ποια είναι η άποψή μου. Εγώ είχα δουλέψει ως συντονίστρια για τις περιφέρειες, προσπαθώντας να δούμε τι στρατηγική έχουν και κάναμε τις αιτήσει τους για τέτοια έργα. Υπάρχει, υπάρχουν πολλές δυνατότητες να βελτιώσουμε την νομοθεσία, να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Και αυτό το χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Γιατί λόγω της κρίσης χρειαζόμαστε δράσεις. Οι δράσεις απαιτούν στρατηγική και συνεργασία. Νομίζω λοιπόν ότι οι εκθέσεις αυτές είναι εξαιρετικά, η έκθεση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και άλλες παρόμοιες. Ο κύριος Ματσάρας. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρκάκη για την έκθεση που υποβάλλει, η οποία έρχεται σε μια πολύ επίκαιρη στιγμή όταν γίνεται έρχεται η αναθεώρηση, η ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Ε, βεβαίως ε, ε, τα προγράμματα αυτά βελτιώνονταν, δεν είχαμε ποτέ ωστόσο αποτελεσματικό αποτελεσματικά επίπεδα. Νομίζω ότι ε, στην αξιολόγηση του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου θα μπορέσουμε να βγούμε μια σειρά νέων ιδεών που θα μπορούσαμε να περιλάβουμε στο 8ο, ούτως ώστε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να βελτιώσουμε την καινοτομία προς όφελος των ΜΜΕ. Αυτό θα πρέπει να είναι μία παρότρινση για την καινοτομία στο μέλλον. Γιατί συχνά λέμε τι καλή που είναι η καινοτομία, τι καλή που είναι η ανανέωση, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε. Και το πρόβλημα δεν αφορά, δεν είναι η έρευνα αυτή καθεαυτή, αλλά η πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στο μέλλον μπορεί να προκύψουν προβλήματα και νομίζω ότι η σωστή προσέγγιση είναι να υπάρχει μία εφαρμογή στις περιφέρειες, αλλά με ε, καταμερισμό στις επιμέρους, σε επιμέρους έργα. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή που θέλει να λάβει το λόγο. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και με την γνωμοδότηση και με το σχέδιο έκθεσης γιατί νομίζω ότι προσεγγίζει ακριβώς την συνολ... έχει ακολουθεί την ίδια συνολική προσέγγιση της Επιτροπής στον τομέα. Δείχνει ότι δουλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση και έχουμε... δίνουμε έμφαση στη συνέργεια. Υπάρχουν κάποια κοινά εργαλεία που οι υπηρεσίες επιτροπή προσπαθούν να δημιουργήσουν από την European Cluster Task Force, από το Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας, τους τρόπους μέτρησης των πολιτικών καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ περιφερειών που υποστηρίζουν διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, το λεγόμενο fast track, ε, ε, η, διαδικασία, η λεγόμενη διαδικασία fast track που ακριβώς αποσκοπεί στην προώθηση ε, τέτοιων μέτρων καινοτομίας. Πολλές δραστηριότητε υπάρχουν. Έχουμε επίσης στο πρόγραμμα μια κοινή ανακοίνωση των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης και, επιχειρήσεων που θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμεινο του 10 με κύριο στόχο την ε, καθοδήγηση των στρατηγικών και των γραμμών των διαφορετικών ταμείων προσαρμόζοντάς τα στις νέες προδιαγραφές και τον νέο προσανατολισμό της πολιτικής 2020. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν οι νέες δυνατότητες συνέργειας και συνεργασίες μεταξύ υποστηρικτών κέντρων αριστείας και προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας μέσω των υπαρχόντων ε, μέσων. Αυτός νομίζω είναι ο στόχος μας και προς την κατεύθυνση εκείνη πηγαίνουμε. Και εμείς σαν επιτροπή και η έκθεση του κυρίου βουλευτή. Επίσης, ε, τέλη Μαρτίου θα εκδοθεί μια στρατηγική έκθεση για την εφαρμογή των διαφθορτικών ταμείων σε σχέση με το νέο πλαίσιο της περίοδου 2007-2013. Θα περιλαμβάνει έκθεση από κάθε κράτος μέλος για την ε, περίοδο προγραμματισμού του πρώτου, της πρώτης φάσης των διαφορετικών ταμείων θα αποτελέσει την ευκαιρία να καταλάβουμε και να δούμε το ξεκίνημα του αντίκτυπου. Είναι νωρί να μιλήσουμε για ένα αντίκτυπο, αλλά το ξεκίνημα του αντικτύπου των μέτρων που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Θέλετε κύριε Χατζημαρκάκη να πείτε κάτι. Εννοείται. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Κομισιόν που μας είπε τι ισχύει αυτή τη στιγμή, αλλά ο κύριος Μετσάρος νομίζω το ανέφερε σωστά. Η βασική έννοια είναι η συνέργεια. Τώρα, τώρα που προγραμματίζεται το πρόγραμμα πλαίσιο 8 και έχουμε νέο επίτροπο που προγραμματίζει νέα πολιτική, που βεβαίω από πλευρά κρατών μελών πρέπει να γίνουν πάρα πολλά όσον αφορά τον έλεγχο του προπολογισμού, τώρα πρέπει να τεθούν ε, οι νέε βάσει. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για το θέμα στρατηγική κατεύθυνση και αν επικεντρωθούμε σε αυτό τον τομέα, δεν ξέρω, ξέρω μάλλον από ποιον ε, με, από ποια περιοχή προέρχεστε και εκεί πέρα πράγματι οι μυαγωγοί παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εκεί πέρα. Γι' αυτό ακριβώς ε, αντιλαμβάνεστε πως χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά για την καινοτομία. Η Σαξονία, παραδείγματο χάρη, είναι υποδειγματική όσον αφορά την οικοδόμηση αυτών των κλάστερ και γνωρίζω πω η Σαξονία στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει αυτά τα περιφερειακά μέσα ακριβώ για να προωθήσει αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση με βάση την καινοτομία για τον συνάδελφο Μπουτικόφερ. Ναι, πράγματι έχει δίκιο. Τελικά πράγματι μιλάμε για μια αϊφόρο, πιο αϊφόρο η οικονομία. Πράγματι πρέπει να, να μπουν εδώ πέρα αυτές οι λέξεις, αυτές οι γνωμοδοτήσεις. Εντάξει, είναι κάπως περιορισμένες, οπότε μπορούν να συμπληρωθούν και από μένα και από τροπολογίες του κυρίου Μπουτικόφερ και Χαίρομαι πράγματι μπορώ ξεκάθαρα να συμπεριλάβω την, την βιομηχανία. Δεν έχω πρόβλημα και με το, το πρασίνισμα της βιομηχανίας που σίγουρα θα προτείνει. Να αναφερθώ όμως σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Λένα Εκ, τι κάνουμε με τα λεφτά. Η Κομισιόν επένεσε το κείμενο, αλλά η Κομισιόν πρέπει να ξέρει πως ε, στο παρελθόν έχουμε κάνει και πάρα πολλά λάθη. Και το βλέπουμε αυτό τώρα στην περίπτωση της Ελλάδας. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε μια χώρα που έχει λάβει πάρα πολλά περιφερειακά κονδύλια στο παρελθόν και μόνο ένα μικρό κομμάτι τους πήγε στην καινοτομία και την έρευνα. Ε, το οποίο όμως ήταν επιτυχές. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε όλη της την, ευρωπαϊκή, την παραγωγικότητα από όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε τώρα πως είναι μια χώρα που ζει μόνο με τις επιδοτήσεις, μόνο με την ε, στήριξη, την τεχνητή αν θέλετε και Βοήθεια. βλέπετε πως πραγματικά αυτός είναι ο μόνος τομέας ο οποίος είναι παραγωγικός στην Ελλάδα. Ε, έχει καταστραφεί οι υπόλοιπε παραγωγικέ δραστηριότητε, υπηρεσίε, τουρισμό έχουν καταστραφεί μέσω τη εσωτερική αγορά. Και βλέπετε τι γίνεται και το πέρα απευθύνομαι κυρίως στα νέα κράτη-μέλη. Χαίρομαι που ο συνάδελφος ε, έλαβε τον λόγο. Ακριβώς που θα ε, μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις ε, συνέργειες μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσουν ειδικά εντό τη ζώνη ευρώ και να μην μπορούν να είναι τόσο παραγωγικέ. Νομίζω το παράδειγμα τη Ελλάδα είναι σαφέ. Πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ προ αυτή την κατεύθυνση Ειδικά μάλιστα τα τα κράτη-μέλη πρέπει να εκπαιδεύσουν αυτούς τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτό το κονδύλι. Αλλιώ δεν έχουν καμία αξία. Το βλέπω στην Ελλάδα από πλευρά ελέγχου του υπερπολογισμού που έχουμε κατάχρηση ή λάθος χρήση των κονδυλίων. Και στο τέλος υπάρχει και αχαριστία. Δείτε τη συζήτηση στην Ελλάδα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Εκεί πέρα πρέπει να ξανασκεφτούμε μήπως πρέπει να αλλάξει ρότα όλη μας η πολιτική. Ε, έφυγε ο κύριος Φανίλης Τελερόη, εν περιπτώσει, αλλά και αυτό συμφωνεί εδώ πέρα μαζί μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα το οποίο ανέφερε και εκείνο. και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, στις προπολογίες τους να πάνε προς αυτή την ε, κατεύθυνση και οπωσδήποτε εγώ θα συμφωνήσω. Σας ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει τον λόγο. Να υπενθυμίσω πως ε, είναι 24 Φεβρουαρίου 12 ε, η ώρα η προθεσμία της τις Σχεδόν, σχεδόν πέρασε δηλαδή. Ναι, συγγνώμη. Ο κύριος Βίνκλερ ζήτησε μία παράταση κατά μία ημέρα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να πάει στις 25. Γιατί πράγματι είναι πολύ σύντομη η προθεσμία και αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω, απευθύνομαι στην γραμματεία εδώ πέρα, 25 όχι 24. Έξυπνη πρόταση, λέει ο Πρόεδρος, Νομίζω ούτω ή άλλως είμαστε πολύ πιεσμένοι. Αν δεν έχει καμία αντίρρηση κανείς. 25 μεσημέρι, 12 η ώρα, ωραία. Έγινε λοιπόν. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί 10 η ώρα έχει οριστεί η ψηφοφορία, εκτός εάν Ω, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Θα ξεκινήσουμε όμως 10 ακριβώς. 10 ακριβώς. Λοιπόν, συνάδελφοι, περνάμε στις ε, ψηφοφορίες, σημείο 7 και τα επόμενα. Εάν μου επιτρέπετε μία παρατήρηση, γιατί είναι κάτι που θα ήθελα και εγώ να τονίσω προσωπικά και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Κοιτάξτε, είναι δύσκολη η ώρα όσον αφορά την τη δουλειά μας και θα έχουμε και άλλες ψηφοφορίες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε, ειδικά όσον αφορά τα, τα έγγραφα, να προετοιμάσουμε την κατάσταση, τα πράγματα έτσι ώστε και οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι εδώ πέρα ή δεν είναι εδώ πέρα στην ώρα τους να μπορούν να διαβάζουν τα έγγραφα. Οπότε συχνά κατατίθενται το προηγούμενο βράδυ συμβιβαστικές ε, τροπολογίες στα, στα γαλλικά. Τέλος Ας αφήσουμε τώρα αυτά όπως έχουν σήμερα για να ψηφίσουμε. Αλλά υποσχέθηκα στους συναδέλφους που μου το είπαν πως θα το πω. Σας παρακαλώ στο μέλλον να προσπαθήσουμε οι συμβιβαστικές ε, τροπολογίες να έρχονται μία μέρα πριν για να μπορούν να τις διαβάσουν όλοι οι συνάλφοι και να είναι τουλάχιστον στα αγγλικά. Γιατί με τις υπόλοιπες γλώσσες είναι και λίγο δύσκολο και δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε και μετά σηκώνεται κάποιο μέσα συνεδρία και λέει θα στο διαβάσω και θα ψηφίσουμε. Οπότε, όσον ακόμα έχουμε χρόνο, ησυχία, οπότε σα το λέω. Τέλο πάντων, σήμερα θα προχωρήσουμε όπω έχουν τα πράγματα, αλλά στο μέλλον θα αλλάξουν. Αυτή ήταν η παρατήρηση. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν τι κάρτε σα να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Μια μικρή δοκιμαστική ψηφοφορία για το εάν στο μέλλον. Τέλος πάντων, δεν, δεν έχει σημασία να, να ψηφίσουμε για το να θέμε ήλιο ή όχι. Δεν θέλετε, Γκέρεκ. Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι φαίνεται έχει χαλάσει η κάρτα. Η δικιά μου δεν ε, λειτουργεί εδώ. Στο ίδιο μηχάνημα οι άλλε ε, λειτουργούν, αλλά η δικιά μου μάλλον έχει χαλάσει. Το δοκίμασα σε οποιοδήποτε μηχάνημα δεν λειτουργεί. Χαλάσει η ίδια η κάρτα. Θα, θα σας μετρήσουμε. Θα σας μετρήσουμε ε, επιπλέον. Λοιπόν, τη ψηφοφορία, Αποτέλεσμα σαφές. 7 δεν μπόρεσαν να, να αποφασίσουν. Θέλω να τους δω. Ποιοι ήταν που δεν μπορούσαν να αποφασίσουν για αυτό το ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Τα μηχανήματα λειτουργούν πλην μια κάρτας που θα πρέπει να προσθεθεί. Πρώτη έκθεση της κυρίας Γκροστέτ. για την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα μέτρα κατά του καρκίνου. Ξεκινάω με την τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ.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 εγκρίνεται με κάποιες ψήφους κατά 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14, 15, 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ψηφίσαμε τη 16. Θέλετε, να ελέγξουμε. Όχι, όχι, ήταν σαφής. Λοιπόν, μια στιγμή, ωραία. Το, το σβήνουμε. Λοιπόν, ε, άρχεται η ψηφοφορία για την 16. Για την 16. 16. Υπάρχει κάποιο παραπάνω από το ΕΛΚ. Κάποιο παραπάνω είναι από το ΕΛΚ. Ποιο Ωραία, πέρας. Αποτέλεσμα, νομίζω ξεκάθαρο. Ευχαριστώ, περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. τρεις παραπάνω από το ΕΛΚ, ακόμη περισσότεροι. Έχουμε θαύματα εδώ πέρα, αυξάνονται και πληθύνονται. Ναι, με συγχωρείτε. Εξακολουθούν να είναι δύο παραπάνω. Δύο από το ΕΛΚ παραπάνω. Ε, ένας παραπάνω είναι τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πέρας της ψηφοφορίας 46 με τρεις αποχές, καμία, καμία Συγχαρητήρια κυρία συνάδελφε και ευχαριστούμε. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Ριέιρα Μαδουρέλ, σημείο 8, διάλογος πανεπιστημίων επιχειρήσεων. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας, ας το ελέγξουμε καλύτερα. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πάλι δύο παραπάνω από το ΕΛΚ. Εντάξει. Πέρας. Αποτέλεσμα, ναι. Ναι, ναι, είναι σαφές. Ναι. Και πρέπει να ψηφίσουμε την 2 τώρα. 2 υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά η 6 καταπίπτει συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 7 καταπίπτει 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 καταπίπτει 13 υπέρ Α, η 13 καταπίπτει επίσης, με συγχωρείτε. Συμβαστική 3, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 καταπίπτει 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18-19 καταπίπτουν 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 23 χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά να ελέγξουμε, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία και πέραση ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα τσίμα τσίμα. Αλλά εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 σε 2 κομμάτια, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε σε τίποτα άλλο, ε. τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική άρχεται ψηφοφορία. Ε, πέρας. Κάποιος είναι παραπάνω από το ΕΛΚ. Ωραία, εντάξει. Πέρας. 48, τρεις αποχές, κανείς κατά. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Οπότε τελειώσαμε και με αυτό. Σημείο 9. Λευκή Βίβλος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πλαίσιο δράσης, κυρία Ματίας, πρέπει να προσέξουμε, να με βοηθήσετε λίγο, γιατί έχουμε τροπολογίες προφορικές. Κυρία Γιόρνταν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας εξηγήσω συντομία το εξή. Στο κατάλογο ψηφοφορίας του ΕΡΚ υπάρχει αρνητικό πρόσημο, όχι γιατί διαφωνούμε με το περιεχόμενο της τροπολογίας, αλλά γιατί κατά τη γνώμη μας τέτοιου είδους δράσεις για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου δεν είναι του θέματος. Θα πρέπει να περιληφθούν σε άλλη έκθεση. Δεν υπάρχει πλέον προφορική τροπολογία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 7 λοιπόν την ψηφοφορία σε τρία μέρη. Πρώτο κομμάτι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά Αχα. απορρίπτεται αποχές απορρίπτεται τρίτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Οχτώ υπέρ κατά να ελέγξουμε. Το 8. Πέρας. Abstimmung geschlossen. Ergebnis. αποτέλεσμα είναι... Der Mann im Computer braucht noch Zeit zum Zählen. Ο άνθρωπος μέσα στο κομπιούτερ χρειάζεται χρόνο για να μετρήσει. Θα ξαναψηφίσουμε λοιπόν το 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Και έληξα. Κάποιο από το είναι παραπάνω. Πέρας. Το αποτέλεσμα. 27 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. 9. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πέρασε. 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Ε, δεκτό. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Δεκτό. 11 υπέρ. Κατά. αποχέ, Δεκτό. 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα του 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αποτέλεσμα. Απορρίπτεται με μία ψήφο περισσότερη. Απορρίπτεται παρόλα αυτά. Απορρίπτεται. Ίσα ίσα. Ναι, ε, κύριο Στουρμες, παρακαλώ. Δεν έχω ακόμα την, ε, την κάρτα μου, οπότε ψηφίζω, τι ψηφίζω, κατά. Υπέρ. Ναι. Ε, είναι αρκετή, είναι παραπάνω η πράσινη, τι γίνεται. Είμαστε τρεις, αλλά λείπει η κάρτα μου. Κατα, κανονικά είμαστε τέσσερις, λέει ο κύριος Τούρμες. Επιτρέπεται να ψηφίσει ο κύριος Τούρμε. Ωραία. Ωραία λοιπόν, άρα εγκρίνεται. Ε, 12 angenommen. Δεκτή. Άρα η 12 περνάμε στην 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά απόχέ δεκτή 18 υπέρ κατά απορρίπτεται 19 υπέρ κατά δεκτή 20 υπέρ κατά δεκτή 21 υπέρ κατά δεκτή ναι 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά 25, 27, 26 καταπίπτουν. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά Να ελέγξουμε. Την 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλα εντάξει. Κάποιος από το ΕΛΚ είναι παραπάνω. Ε, είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Κατά... Όχι, ναι, συγγνώμη, ναι. Πέρας ψηφοφορίας ενός. Εγκρίνεται με 31, αντί 22. 5 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε. Την 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μια στιγμή. Ναι, απορρίπτεται. Συν ο κύριο Γκύρη καρά 27 κατά. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε τις ψηφοφορίας. Ναι. Εγκρίνεται συγχαρητήρια και ευχαριστούμε. Περνάμε σημείο 11. Η φόρο μέλλον για τις μεταφορές. Κάντσιαν. Α, συγγνώμη, στο 10 είμαστε. Γεωργία. Γεωργία. Λοιπόν, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Πιο αργά, πιο αργά. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη 2 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 3 σε 4 κομμάτια. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τρίτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέταρτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 σημείο α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9, 8, 7, 5 καταπίπτουν. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10, 11, 12, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά α, αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 17 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 18 υπέρ Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 σε δύο κομμάτια υπέρ του πρώτου. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 σε δύο μέρη, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην τελική ψηφοφορία Αρχική ψηφοφορία πέρας ένας παραπάνω από το ΕΛΚ εντάξει πέρας 45 υπέρ, ένας κατά 5 αποχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Επόμενη, 11. Αντώνιο Καντσιάν. Μέλλον για τις μεταφορές. Έχετε τον κατάλογο. Περνάμε σημείο 1 υπέρ, κατά αποχές. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 1. Έρχεται η σωφορία. Πέρασε. Πέρασε. Δεκτή. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρία. Καταπέμπτη. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατά πίπτουν 7 έως 13 και περνάμε σε 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 15 κατά πίπτη 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ Α, τι ψηφίσαμε ήδη, με συγχωρείτε, ναι. 18, ε, άρα 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21, 22, 23, 24 καταπίπτουν. 25 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε το δεύτερο κομμάτι αρχιετή ψηφοφορία ένας παραπάνω από το ΕΛΚ πέρας απορρίπτεται ναι ναι απορρίπτεται απορρίπτεται απορρίπτεται παρόλα αυτά γιατί έχουμε ισοψηφία 26 υπέρ κατά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 πρώτο τμήμα της 42 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. Α, ναι, ναι. Εντάξει, άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, οπότε... Με πρώτο τμήμα καταπίπτει. Οπότε, ξανά. 42 το πρώτο τμήμα καταπίπτει, άρα ψηφίζουμε το υπόλοιπο. Οπότε, παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τούρμες και επί της διαδικασίας την 33 ε, την ψηφίσαμε παρά το ότι έπρεπε να έχει καταπέσει εάν περάσει 37. Ναι, ε, ε, πώς μπορείτε να το ελέγξετε. Δεν ψηφίσαμε την... είχε απορριφθεί ή 37. Ωραία, λοιπόν, τελική ψηφοφορία υπέρ... Ε, άρχιτη ψηφοφορία μάλλον, με συγχωρείτε. Ε, ναι, όχι. Πέρα, με συγχωρείτε. Ένα Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ, όπω πάντα. Ε, είναι πάρα πολύ εδώ μέσα. Πέρα. 46, μια αποχή, τρεις κατά, συγχαρητήρια, ευχαριστώ. Και με αυτό τελειώσαμε. Οπότε τελειώσαμε εγκαίρως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε να συνεχίσουμε την ημερήσια διάταξη. Και περνάμε σημείο 12. Το οποίο... Όσοι θέλετε να φύγετε παρακαλώ φύγετε σύντομα και χωρίς ε, ε πολυφασαρία για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Το κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική θάλασσα. Η συνάδελφος κυρία Εκ είναι η συγγήτρια και της δίνω πάρα αυτά το λόγο. Ε, λέω πάρα αυτά, αλλά καλό θα ήταν περιμένουμε ένα λεπτουδάκι γιατί παραγίνεται φασαρία στην αίθουσα. Παρακαλώ, φύγετε όσοι θέλετε να φύγετε, όσοι ήρθατε να ψηφίσετε να φύγετε γρήγορα και να μην κάνετε πολύ φασαρία αν γίνεται. ούτως ώστε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση του επόμενου θέματος στην ημερήσια διάταξη. Συνάδελφοι, η κυρία Εκ έχει το λόγο μόνο, μόνη της. Όλοι οι άλλοι σταματάτε να μιλάτε. Thank you, Uh, uh, Θα περιμένω, Πρόεδρε, για να μπει λίγη τάξη Σάρ. Wir würden gerne weitermachen. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, θέλουμε να συνεχίσουμε. Um, Ευχαριστώ. Όταν υιοθετήθηκε το κοινό πρόγραμμα, όταν μπήκε στην ημερήσια διάταξη το κοινό πρόγραμμα έρευνα και ανάπτυξη βαλιστική θάλασσα την περασμένη φορά, ήθελα να υποβάλω, να περάσω μια σειρά σημαντικών επιχειρημάτων υπέρ του προγράμματος αυτού. Όλοι ξέρουμε την σοβαρή κατάσταση της Βαλτικής. Όλοι γνωρίζετε το ιστορικό των πολύ σημαντικών ε, ισχυρών αποφάσεων του Συμβουλίου για την Βαλτική. Να τονίσω πόσο την απόλυτη υποστήριξη των δύο επιτρόπων, της Επιτρόπου για το Περιβάλλον και του Επιτρόπου Έρευνας, για το πρόγραμμα αυτό, Ωστόσο συνεχίζω να έχω ορισμένε ανησυχίες που βασίζονται στην πρόταση της Επιτροπής. Όχι στο περιεχόμενο, το εξαιρετικό περιεχόμενο του προγράμματος Bonus 169, αλλά στην ύπαρξη προσπαθειών να δυσκολέψουν την κατάσταση. Παρότι δηλαδή και το Συμβούλιο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θέλουν να διευκολύνουν την διαδικασία, υπάρχουν στην έκθεση Επιτροπής κάποια κομμάτια που είναι προβληματικά. Η συζήτηση δεν αφορούσε το κατά πόσο κάποια σημεία θα ανήκαν ή όχι στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο ή στο αν το πόνους ε, πρέπει να υπάρχει όχι, αλλά στα νέα στοιχεία που παρουσιάζονται, που είναι αποτέλεσμα και συνέπεια του προγράμματος δύο φάσεων, με ένα στρατηγικό τμήμα και ένα ερευνητικό τμήμα. Υπάρχουν ήδη έργα του 169 που λειτουργούν, που δουλεύουν. Η πρόταση της Επιτροπής λοιπόν για μια ε, δίχρονη προσέγγιση σε δύο χρόνους είναι καινοτομία, αλλά οι ερευνητές που μετέχουν ήδη σε έργα στα κράτη-μέλη συμφώνησαν να δουλέψουν με τη στρατηγική αυτή, όπως θέλει η Επιτροπή, και κατόπιν να προχωρήσουν στην πλήρη ολοκληρωμένη περίοδο έρευνας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για να προσελκύσουμε τους καλύτερους, καλύτερους ερευνητές το πέρασμα από την πρώτη στη δεύτερη φάση να μην δυσχεραίνεται αλλά αντίθετα να γίνεται όσο πιο εύκολο μπορούμε. Διότι η εισαγωγή νέων στοιχείων έτσι όπως γίνονται τα ερευνητικά έργα είναι ελπιδοφόρο, είναι καλό, αλλά δεν πρέπει να, είναι, να, να γίνεται εργαλείο ε, τροχοπέδι στο έργο. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Κάτι άλλο. Χρηματοδότηση. Και εδώ μπαίνει ένα κενό, αυτό που, ένα καινούριο στοιχείο, αυτό που λέμε κοινό κορβανάς. Το είχαμε πει στην προηγούμενη συνάντηση. Και αυτό είναι νέο στοιχείο. Πολλά ερευνητικά προγράμματα προσπαθούν να δουλέψουν όσο καλύτερα γίνεται σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο σε 8 χρόνια θα υπάρχει μεγαλύτερη νομοθετική προσέγγιση για ένα μια ολοκληρωμένη αρχή κοινού κορβανά. Ωστόσο τώρα τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν προβλήματα με την ε, δική τους νομοθεσία και συνταγματικού χαρακτήρα. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα θεωρητικό ε, κοινό κορβανά, την ιδέα δηλαδή ενσωμάτωσης μόνο της διαχείρισης των οικονομικών των χρηματοοικονομικών διαστάσεων, αλλά να λάβουμε υπόψη τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη-μέλη, Γερμανία, μικρά κράτη-μέλη. Μεγάλες δυσκολίες λόγω του κόστους. Αυτό είναι δεύτερο πρόβλημα. Στην έκθεση μου προσπαθώ να το καλύψω αυτό. Θέλω να βλέπω πώς έχουν τα πράγματα στο μέλλον, να λάβω υπόψη μου τα σχόλια από την προηγούμενη συζήτηση και να καλύψω και όσο καλύτερα γίνεται και την διάσταση της συνεργασίας με τη Ρωσία. Ξέρουμε ότι η Ρωσία επηρεάζει σημαντικά την κατάσταση στη Βαλτική και θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να μας προσφέρει, να μας προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης και άριστης συνεργασίας με Ρώσους ερευνητές. Και εδώ θέλουμε κάποια δουλειά για να τους ενσωματώσουμε πλήρως στο πρόγραμμα, αλλά ήδη και στο πρώτο πρόγραμμα Bonus In έχει ξεκινήσει συνεργασία με τη Ρωσία, δουλεύει σε διμερή επίπεδο, σε διμερές επίπεδο. Δηλαδή, μέλη του Bonus In συνεργάζονται με τη Ρωσία. Και στο πρόγραμμα μετέχουν ερευνητές Ρώσοι, πηγαίνουν σε σεμινάρια, προσπαθούν να βρουν κοινό πεδίο συνεννόησης. Όπως σας είπα, το bonus in, υπάρχουν προγράμματα bonus in που, που έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν με θετικά αποτελέσματα, πολύ θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Έγινε πριν από δύο εβδομάδες μόνο μια μεγάλη σύνοδος κορυφής για την κατάσταση στη Βαλτική παρουσιάστηκαν τα επιστημονικά ευρήματα παρόντων των αρχηγών κρατών. Πολλά από τα ευρήματα προέρχονταν από έρευνες του Bonus -in. Τι χρειαζόμαστε τώρα, χρειαζόμαστε μια γρήγορη απόφαση για τον Bonus 169. Γρήγορα. Και γιατί γρήγορα, διότι η κατάσταση στη Βαλτική είναι πολύ δύσκολα, δύσκολη περιβαλλοντικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν να, έχουμε, να προχωρήσει η επιστημονική έρευνα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κυρίως διότι αν υπάρξει μια χρονική απόκληση μεταξύ του τι γίνεται τώρα και του bonus 169 που είναι και πιο διευρυμένο και πιο στρατηγικά στοχοθετημένο, θα μπορέσουμε να έχουμε μια απάντηση όχι μόνο για το πώς είναι η κατάσταση, αλλά και γιατί έγινε η κατάσταση έτσι όπως έγινε και επιπλέον θα έχουμε και κάποιες λύσεις. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ τα μέλη για την συμμετοχή στο, στην επεξεργασία των ε, τροπολογιών και ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση. Οι συνάδελφοι τώρα έχουν το λόγο. Πρώτα ο κύριος Γκέρεκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μερικές γενικές παρατηρήσεις. Ο προτινόμενος κανονισμός για την κατάσταση στη Βαλτική περιλαμβάνει κάποια πολύ σοβαρά στοιχεία. Μία ανάγκη ε, στρατηγικού προγραμματισμού. Χωρίς ε, αυτή την ε, φάση δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ποιοτικά αποτελέσματα. Από ό,τι ξέρω πρόκειται για ένα ευρύ σχέδιο δράσης και μια ευρύτερη στρατηγική που δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τη θάλασσα, τη Βαλτική θάλασσα, αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα. Στο σημείο 6.2 ε, περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μου το εκθέσει. Και επίσης έχουμε το άρθρο 4 για το κοινό ερευνητικό κέντρο. Περί τίνος πρόκειται, γιατί Πολύ ακροθυγώ αναφέρονται τα σημεία αυτά στα συμπεράσματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των νέων χωρών μελών στην ε, Βαλτική θάλασσα χρήση διαφορετικής προσέγγισης. Καταρχήν ε, το ερευνητικό δυναμικό είναι πολύ διαφοροποιημένο μεταξύ των συμμετοχών των χωρών και ε, χρειάζεται ένα καλύτερο πλαίσιο γιατί μπορεί να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό αλλά δεν υπάρχει εξοπλισμός ούτε αρκετά εργαστηριακός εξοπλισμός. Υπάρχει μεγάλη στέρηση σε αυτό το θέμα των ε, εργαστηρίων. Αυτές, αυτοί οι περιορισμοί θα πρέπει να αρθούν κατά τη γνώμη μου. Γιατί πρόκειται για πολυγονικές, όπως λέμε, μελέτες και έρευνες που θα γίνουν επιτόπου στο οικοσύστημα της Βαλτικής. Επίσης, ε, πολλές χώρες ε, δεν μπορούν να δεχτούν αυτό το κοινό κορβανά, το κοινό ταμείο. Και από νομική άποψη είναι απαράδεκτη αυτή η πρόταση, αλλά και από άποψη ε, δυνατότητας υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων. Τώρα, για τη στρατηγική φάση. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα. Δεν πρέπει να περιορίσουμε τη διετία που προτείνεται. Και για να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις. Στην στρατηγική αυτή φάση θα πρέπει να προσδιοριστούν κάποιες ερευνητικές προτεραιότητες για το σύνολο της Βαλτικής θάλασσας και των οχθών της. Επίσης θα πρέπει, εκτός από τις προτεραιότητες, να γίνουν και κάποιες ε, προετοιμασίες επενδυτικού χαρακτήρα για τις έρευνες αυτές. Θα πρέπει να δημιουργηθούν πραγματικά ερευνητικά εργαστήρια για αυτές τις πολυγονικές έρευνες και τις εργαστηριακές μελέτες. Και όταν μιλώ για ερευνητικά εργαστήρια, έχω υπόψη μου κυρίως ε, τις νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές δηλαδή προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004. Οι χώρες αυτές έχουν πλούσια εμπειρία, έχουν καλό πλαίσιο, αλλά δυστυχώς ε, στερούνται τεχνικών εξοπλισμών στα εργαστήριά τους, στα ερευνητικά τους εργαστήρια. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χάση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για την ε, πολύ αξιόλογη έκθεσή της και να συμφωνήσω με την προσέγγισή της, γιατί συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ε, στο πρόγραμμα αυτό και να βρούμε έναν τρόπο για να επιταχύνουμε τις εργασίες και να μην περιμένουμε πολύ μέχρι να θέσουμε σε, σε κίνηση αυτό το νέο μπόνους. Το νέο μπόνους αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ καλό και στηρίζεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βαλτική θάλασσα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βαλτική θάλασσα είναι πρωτοβουλία που εκπορεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα η Σουηδική Προεδρία δραστηριοποιήθηκε ενεργά για την πρόθεση αυτής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βαλτική. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει σημαντική διάσταση απόψεων ή διαφορές ε, ως προς το περιεχόμενο. Ίσως ε, υπάρχει ένα διαδικαστικό ζήτημα που το επισήμανε η συγγήτρια για αυτό το θέμα του κοινού ταμείου, του πραγματικού εικονικού κοινού ταμείου. Υπάρχει πρόβλημα σε ορισμένες χώρες γιατί δεν υπάρχουν νομικές βάσεις για τη σύσταση ενός τέτοιου κοινού κορβανά. Δεν ξέρω αν ε, ευσταθούν τα νομικά επιχειρήματα που επικαλούνται ορισμένε χώρες για να απορρίψουν την πρόταση για το κοινό ταμείο, θα πρέπει να το ελέγξουμε και να βρούμε πρώτα απ' όλα μια πρακτική λύση για να κινητοποιήσουμε τον πόνους. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινού κανόνες ε, χρηματοδότησης και διαδικασίες, ιδιαίτερα όταν καταλήξουμε στην πρόταση του κοινού προπολογισμού του κοινού ταμείου. Για να μην περιπλέξουμε την εφαρμογή του συστήματος εφόσον θα έχουμε ορισμένε χώρε που θα εφαρμόζουν του κοινού κανόνε και άλλε που θα εφαρμόζουν την εθνική του νομοθεσία. Γιατί κάθε εθνική νομοθεσία έχει ιδιαιτερότητε για τέτοια θέματα. Ελπίζω να επιταχύνουμε τη διαδικασία παρά την πρόταση για το κοινό ταμείο, τον κοινό προϋπολογισμό. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θα συζητήσει σήμερα το πρωί και αυτή τη γνωμοδότησή της και κατά πάσα πιθανότητα να υποβάλει, θα υποβάλει προτάσεις που θα ενισχύουν τις περιβαλλοντικές πτυχές της έκθεσης. Ευελπιστώ ότι και η δική μας Επιτροπή θα λάβει υπόψη την ε, θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Βαλτική θάλασσα είναι από τις πιο μολυσμένες θάλασσες του κόσμου. Πολλοί βέβαια πιστεύουν ότι στη Βόρεια Ευρώπη η οργάνωση είναι άψογη, όλοι σέβονται την νομοθεσία, η προστασία του περιβάλλοντος ε, είναι ύψιστη προτεραιότητα. Όλα είναι ρόδινα στις σκανδιναβικές χώρες. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι η Βαλτική θάλασσα είναι από τις πιο μολυσμένες θάλασσες του κόσμου. Άλλωστε πρόκειται για μια εσωτερική πια θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισημαίνει στην έκθεσή της και η αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση του οικοσυστήματος Βαλτικής. Κύριος Μπαλτσίτης, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για μια πληρέστατη έκθεση που αντικατοπτρίζει και τις συζητήσεις που είχαμε στην Επιτροπή μας. Να Κάνω κάποια σχόλια, ωστόσο. Χρηματοδότηση. Η τροπολογία 19 παρέχει τη δυνατότητα εικονικού κοινού ταμείου. Πρόκειται για μια πρακτική πρόταση. Ωστόσο, Πιστεύω ότι στην τροπολογία πρέπει να φύγει η φράση που λέει δικαιολογημένες περιπτώσεις. Υπάρχει επίσης μία τροπολογία για το ρόλο της Επιτροπής και την αξιολόγηση, στην αξιολόγηση της Κομισιόν. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική ή καθυστερήσει υπερβολικά. Μπορεί το πρόγραμμα ολόκληρο να καθυστερήσει. Δεν λέμε ότι, γιατί λέμε ότι η Επιτροπή μπορεί, να, μπορεί δύναται να συμβάλλει, αλλά ε, αυτό συμβαίνει σε δικαιολογημένε περιπτώσει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι προφανές ότι το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται και αφορά στις χώρες της Βαλτικής. Άρα η συνεργασία με την ρωσική πλευρά είναι αναπόφευκτη και αναπόδραστη. Η, η υπερβολικά ανοιχτή όμως αναφορά στην, ε, στο κείμενο αυτό σε, στη Ρωσική Ομοσπονδία δίνει, κανείς την, δίνει σε κάποιον την εντύπωση ότι δεν πρόκειται πια για πρωτοβουλία κρατών της Ένωσης αλλά για μια πρωτοβουλία ενός ευρύτερου αριθμού κρατών. Απλά να πούμε ότι καλωσορούμε, προσκαλούμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να μετάσχει, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Οντινό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Εξαιρετική δουλειά έκανε. Τρεις βασικές παρατηρήσεις για την έκθεση. Συντονισμός, των οχτώ επιστημονικών κοινοτήτων των κρατών μελών που μετέχουν στο πρόγραμμα με συμμετοχή της Ένωσης. Μήπως θα έπρεπε να προβλέψουμε ότι η Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό πέραν των 8 κρατών μελών, θυμάμαι κάτι συζητήσει που είχαμε στο παρελθόν για το σχέδιο Ευρώπη Μεσόγειος, όπου αφού είπαμε ότι ενδιαφέρει τα κράτη, τα παράκτια κράτη της Μεσογείου, ενδιαφέρει και την Ένωση. Μήπως λοιπόν θα πρέπει και εδώ να πούμε ότι η Ένωση εμφανίζεται ως μετέχον πέραν και ε, επιπλέον των κρατών μελών. Επίσης, μου κάνει εντύπωση, μιλήσαμε για την Ρωσία, αλλά δεν περιλαμβάνεται πουθενά, δεν γίνεται πουθενά μνήμα της Νορβηγίας. Είναι μέλος του ΕΟΧ. Προφανώς δεν βλέπουν στη Βαλτική, αλλά αν συγκρίνουμε και με το ευρωμεσογειακό σχέδιο, είχαμε συμπεριλάβει εκεί την Πορτογαλία και τη Μαυριτανία. Παρότι δεν βρέχονταν από τη Μεσόγειο. Μήπως με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την Νορβηγία με ρητιμνία. Κάτι ακόμα. Ε, δεν είδα προσεκτικά την οικονομική διάσταση. Ωστόσο, ε, τα προγράμματα έρευνας έχουν τόσο περίπλοκο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα έπρεπε να τροποποιηθεί. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή μήπω θα έπρεπε να εξετάσει την απλούστευση της διαδικασίας. Δεν πρέπει η επιστημονική κοινότητα να ε, ε φορτώνεται με τόσο περίπλοκα διοικητικά ζητήματα. Ευχαριστούμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ θερμά την εισηγήτρια για την πολύ αξιόλογη της έκθεση και να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές για την συμβολή τους στη συζήτηση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εν συνδομία τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορισμένα κέρια τμήματα της συζήτησης. Το πρώτο σημείο αφορά τη στρατηγική φάση του προγράμματος. Η στρατηγική φάση του προγράμματος ε, είναι πολύ σημαντική όπως ε, υπογράμμισε και η συγγήτρια γιατί θα πρέπει να καθοριστεί το στρατηγικό ερευνητικό πρόγραμμα και θα πρέπει σε αυτή τη στρατηγική φάση για αυτή τη στρατηγική φάση να προβλέψουμε επαρκή χρόνο, μία αρκετά μεγάλη προθεσμία, ώστε να μπορέσει το επιτελείο του μπόνους να ανταπεξέλθει στο περίπλοκο και πολύ σημαντικό καθήκον και έργο που έχει. Δεν είμαι υπέρ της σύντμησης του χρόνου της στρατηγικής φάσης, γιατί μια τέτοια περικοπή του χρόνου θα αποβεί εις βάρος της ποιότητας της πρωτοβουλίας αυτής. Επίσης επιμένω ότι η στρατηγική φάση δεν είναι μια διαδικασία αν θα γίνει δεν θα γίνει το πρόγραμμα. Είναι μια φάση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει το επιτελείο του Μπόνους να καθορίσει το στρατηγικό ερευνητικό πρόγραμμα και θα υπάρξει μια συνέχεια μεταξύ της στρατηγικής φάσης και της ε, φάσης ε, θέσης ε, σε εφαρμογή του προγράμματος. Και το θέμα του τρόπου χρηματοδότησης, το θέμα του κοινού ταμείου του κοινού Καρβανά είναι πολύ σημαντικό και εδώ θα πρέπει να επαναλάβω την αποκρισταλωμένη άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και την επιμονή της στην πρόταση του Κοινού Ταμείου. Μην ξεχνάτε και την έκθεση Βαμβέλσεν. Εκεί επισημαίνεται ότι το θέμα του Κοινού Ταμείου είναι θέμα ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης ουσιαστικά. Και το Κοινό Ταμείο είναι ο απλούστερος τρόπος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της πρωτοβουλίας αυτής. Το Κοινό Ταμείο επίσης ε, δίνει τα εχέγγυα στις ε, ερευνητικές ομάδες ότι θα χρηματοδοτηθούν. Και μάλιστα ιδιαίτερε ερευνητικές ομάδες των χωρών που θα ε, χρηματοδοτήσουν με μετρητά τις ε, ερευνητικές προσπάθειες. Και επειδή τα μετρητά θα είναι λίγα. Είμαστε υπέρ της πρότασης του κοινού ταμείου. Είναι το εχέγγυο για την χρηματοδότηση των ε, ερευνητικών προσπαθειών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς πόρους και τις υποδομές. Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν είναι να περιορίσει, να περικόψει το ρόλο των υποδομών ή να συρρυκνώσει την ποσότητα ή την ποιότητα των ερευνητικών υποδομών που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα αναζήτησης ισορροπίας μεταξύ των συνεισφορών που θα γίνουν υπό τη μορφή των υποδομών και των συνεισφορών υπό την ε, μορφή των μετρητών ή των οικονομικών πόρων. Σίγουρα οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές, αλλά χρειάζεται μια σωστή αναλογία μεταξύ των συνεισφορών που γίνονται στις υποδομές και των ε, συνεισφορών που γίνονται της μετρητής. Γιατί πρέπει να αμυφθούν οι ερευνητές να χρηματοδοτηθούν τα ερευνητικά προγράμματα. Σε ό,τι αφορά την παρουσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα για την πλήρη συμμετοχή της Ρωσίας στην πρωτοβουλία αυτή, αλλά και στο παρελθόν ε, κατέστη δυνατό κάτι τέτοιο. Η Ρωσία μπορεί να συμμετέχει με βάση του κανόνε που ισχύουν στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. γιατί την Νορβηγία είναι κάπω διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ήδη υπάρχει συμφωνία σύνδεση με τη χώρα αυτή. Οπότε η συμμετοχή των νορβηγικών ε, ερευνητικών ομάδων είναι εφικτή. Με αυτή τη λογική και το πρίσμα θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και με τελείως επικοδομητικό πνεύμα θα λάβουμε υπόψη τις απόψεις και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω πως ε, θέλει εδώ πέρα τον λόγο ξανά η κυρία εισηγήτρια. Yeah. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια, την παρα... τις παρατηρήσεις και την υποστήριξη που εξέφρασαν. Συμφωνώ με τα σχόλιά σας και συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Άλλωστε θα έχουμε τους σκιώδεις ηγετές και τους άλλους ενδιαφερόμενους ε, και άλλες συναντήσεις προκειμένου να συμπεριλάβω τις παρατηρήσεις τους. Και για την Ορβηγία συμφωνώ. Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο ώστε ένα τέτοιο σχέδιο που ισχύει για τη Μεσόγειο να ισχύσει παρόμοιο για τη Βαλτική και να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ή να είναι αποτελεσματικά και στοχοθετημένα. Η Νορβηγία έχει πολύ καλή έρευνα για το θαλάσσιο περιβάλλον, υψηλού επίπεδου και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και τη δική της συμμετοχή. Αλλά μέχρι στιγμής η ίδια η Νορβηγία έχει προτιμήσει να μην συμμετέχει σε αυτή την ε, πρωτοβουλία. Και μάλιστα περιμένω το απόγευμα ε, μία αντιπροσωπή από την Νορβηγική Βουλή ε, σίγουρα θα τους θέσω αυτό το ζήτημα. Τώρα, για τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτιμώ ιδιαίτερος την προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα σχόλιά της και μετά από αυτά που μας είπε ο κύριος Μάτι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στο κείμενο και να τα έχουμε υπόψη και για, τις, ε, για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων ότι η απόφαση για τη δεύτερη φάση από τη, από τη μετάβαση στρατηγική στην εφαρμοστική δεν είναι μία απόφαση go-no-go, no go, ένα είδους ε, check-up, διαγνωστικού ελέγχου. Και καλό είναι αυτό να το κατοχυρώσουμε και γραπτός, γιατί η επιστημονική κοινότητα είναι πολύ απαιτητική και πολύ άριθμη και θέλουμε να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή της και την πλήρη αφοσίωσή της στο πρόγραμμα. Γι' αυτό καλό είναι να τους καθησυχάσουμε. Για το κοινό ταμείο, τον κοινό κορβανά, είναι κάτι που προτάθηκε στη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος και κάτι τέτοιο δημιουργεί δυσκολίες, γιατί τα κράτη-μέλη δεν πρόλαβαν να τροποποιήσουν την ομοθεσία τους. Ελπίζουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο με το 8ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο, όταν ε, υποβληθεί και θα υπάρξει περιθώριο κάποιε διετία για την προσαρμογή. Θα πρέπει όμω να αξιοποιήσουμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα, γιατί θέλουμε όλα τα συμμετέχοντα κράτη να παραμείνουν εντός του προγράμματο. και να καταβάλουν τις, ε, όλες τις προσπάθειες που χρειάζονται. Και συμφωνώ με την κυρία Χάση ότι η κατάσταση είναι σοβαρή. Όταν συζητούμε το θέμα με τη Γερμανία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συμμετοχή και της Γερμανίας και να βρούμε μια διατύπωση που θα ικανοποιεί και τη Γερμανία. και ίσως ε, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ένα εικονικό ε, κοινό, ταμείο που προϋποθέτει μία συμφωνία επί της αρχής και προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, αλλά ταυτόχρονα θα εφαρμόζει την επικουρικότητα. Και αυτό ε, είχε λυθεί με τα πρώτα τρία προγράμματα του Bonus 169. Πιστεύω ότι θα ισχύσει και για το τέταρτο πρόγραμμα του Bonus 169. Και βλέπω ότι ε, ναι, θετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τις συνεισφορές σε υποδομές και σε είδος ε, της μετρητής. Αυτές είναι οι διαφορές που υπάρχουν και τις γνωρίζουμε μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών και εδώ θα, θα πρέπει να αφήσουμε προσπαθειών για να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες υποδομές και να εξασφαλίσουμε και τα μετρητά όπου χρειάζονται. Και χρειαζόμαστε εδώ την ε, στερεότυπη διαδικασία που ισχύει για όλα τα ερευνητικά προγράμματα σε ό,τι αφορά τι συνεισφορέ σε είδο και με μετρητά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια βάση και για το, την πρωτοβουλία bonus. Τέλος, για τη Ρωσία, ναι, όντως υπάρχουν δυσκολίες, Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει σε μια συνολική συμφωνία με τη Ρωσία που θα καλύπτει και άλλους τομείς και όχι μόνο την ε, έρευνα και την, τον πολιτισμό αλλά και την ενέργεια που είναι θέμα μείζωνος σημασίας για την Επιτροπή μας. Στην τελευταία διάσκεψη κορυφής του Μπόνους που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στο Ελσίνκι είδαμε ότι η Ρωσία τη χρησιμοποιήσει ως ευκαιρία για συμμετοχή και συζήτηση. Και μάλιστα έγιναν κάποιες υποσχέσεις, δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις από τη ρωσική πλευρά στην διάσκεψη αυτή κορυφής του Ελσίνκη. Θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στο σχέδιο μπόνους και νομίζω ότι είναι μια καλή αφετηρία και για το μέλλον, για τις μελλοντικές εξέλιξεις. Έχουμε και το χρονοδιάγραμμα και με την αμέριστη υποστήριξη και της Ισπανικής Προεδρίας θα προχωρήσουμε ολοταχώς. Η Ισπανική Προεδρία δήλωσε ότι θα συμπεριλάβει αυτό το θέμα στο, ερευνητικό, στο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνα την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω, ευελπιστώ μάλλον, ότι το θέμα αυτό θα περάσει στην Ολομέλεια του Ιούνιου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 3 Μαρτίου μέχρι τις 3 Μαρτίου τροπολογίες. Τελειώσαμε και με αυτό το σημείο, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο 13 πράσινη βίβλιο της Κομισιόν για τα βιολογικά απόβλητα. Εδώ πέρα τον λόγο έχει ο κύριος Τζάιλς Τσίτσεστερ, ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω πως δεν είναι, πως είναι τυχαίο το ότι είναι το σημείο 13 στη Μέση Διάταξη, γιατί Πιστεύω ότι το 13 θα μας φέρει τύχη για το θέμα που με απασχολεί, όχι ατυχία. Είναι η γνωμοδότηση που στέλνουμε προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την πράσινη βίβλο, για την ακίνηση Επιτροπής σχετικά με την διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων. Μεταξύ των προτάσεων που έχω συμπεριλάβει, δίνουμε έμφαση στις δικές μας αρμοδιότητες την, το δυναμικό παραγωγής ενέργειας από τα βιολογικά απόβλητα. Και εκεί εστιάζει την ε, σημασία της, ε, την δίνει έμφαση η γνωμοδότηση. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι να ενθαρρύνουμε τη χρήση αυτού του πόρου για την παραγωγή ενέργειας σαν τμήμα της συνολικής πορείας της Ένωσης προς την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, με στόχο και την ενίσχυση της ε, ασφάλειας στην τροφοδοσία ενέργεια, γιατί προφανώς η βιομάζα είναι εσωτερική παραγωγή. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ιδιαίτερα επίμαχο στη γνωμοδότηση. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη των συναδέλφων, αν έχουν κάποια. Ελπίζω πάντως ότι αυτά που καταθέτουμε εδώ θα περάσουν στους φίλους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αν θα μπορούσα να υπογραμμίσω δύο σημεία που θεωρώ σημαντικότερα, θα ήταν τα σημεία 7 και 8 κατά την Το σημείο 7 υπογραμμίζει την δυνατότητα πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, ενώ το 8 τονίζει τη σπουδαιότητα του να κρατήσουμε όλες τις τεχνολογικές επιλογές ανοιχτές. Είναι ένας τομέας ε, όπου υπάρχει, που υπάρχει ακόμα υπάρχουν ακόμα μεγάλες δυνατότητες και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτά, πρόεδρε. Από πλευράς μου σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φαν Βρέμπτ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την γνωμοδότηση αυτή που έχει σημαντικά στοιχεία μπορούμε οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε αλλά σε κάποια σημεία βεβαίω ε, πρέπει να δούμε την γνωμοδότηση της, ε, της ε, Επιτροπής μας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος την οποία πρέπει να ενισχύσουμε. Το πρώτο κομμάτι αφορά το όραμα για το ποια πρέπει να είναι η ιεραρχία των αποβλήτων. Ε, ξέρετε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάμε στην πρόληψη, μετά επαναχρημοποίηση, επαναξιμοποίηση και ανακύκλωση, μετά ε, παραγωγή ενέργειας και τέλος η χωματερή όσον αφορά τα βιοαπόβλητα. Αυτό σημαίνει πως σε πολλά κράτη-μέλη πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσουμε για να γίνει πολύ καλύτερη συλλογή για λαχανικά, φρούτα, δημητριακά και για απόβλητα παραγωγής τροφίμων ε, και να υπάρξει και ένας διαχωρισμός ε, της ποιότητας για το τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ και ω λείπασμα και για να καταπολεμηθεί η διάβρωση του εδάφους και τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κομπόστ και για βιοαέρια. Νομίζω μια τέτοια συμπλήρωση είναι πάρα πολύ σημαντική και στηρίζει το όραμα του εισηγητή για την ανάκτηση της ενέργειας. Δεύτερον, που μάλλον δεν θα συμφωνεί τόσο πολύ ο εισηγητής. Εγώ νομίζω πως πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιό να επεξεργαστεί συγκεκριμένα οδηγία για τα απόβλητα και νομίζω πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάμε σε μεγαλύτερη δυνατή χρήση του πιθανού αυτού δυνητικού αποθέματος και χρειαζόμαστε ένα ξεχωριστό όραμα με μια ξεχωριστή οδηγία, με ξεχωριστούς στόχους για τα απόβλητα και είναι αυτό σημαντικό και για τους στόχους και για να έχουμε ίσο ανταγωνισμό. Υπάρχουν κράτη-μέλη που κάνουν μεγάλες επενδύσεις για την ανάκτηση και την επεξεργασία και νομίζω πως μπορεί να τη στηρίξει αυτές τις επενδύσεις μια τέτοια οδηγία. Μια οδηγία μπορεί να συνεισφέρει στην, στον ίσο ανταγωνισμό, όπως είπα, στο δίκαιο ανταγωνισμό και για τα νέα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν πω δεν θα επιτευχθεί αυτό ο στόχο με συμπλήρωση τη υπάρχουσας τη γενική οδηγία για τα απόβλητα. Οπότε μια ιδέα που προτείνω εγώ είναι έκκληση στην Κομισιόν για το ότι χρειάζεται μια ξεχωριστή οδηγία. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Έχετε το λόγο. Υπάρχει κάποιο που θέλει να μιλήσει. Ορίστε. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε κι εμείς ε, να πούμε. Ε, η ιεραρχία των αποβλήτων ε, ρυθμίζεται στην οδηγία πλαίσιο και προφανώς η αντίδραση στην οδηγία είναι η πρώτη δράση, μετά ανακύκλωση, μετά ανάκτηση και εν τέλει η ταφή. Αυτό επικυρώθηκε πρόσφατα στην νέα οδηγία πλαίσιο, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Για το δεύτερο θέμα, αν χρειάζεται δηλαδή ειδική οδηγία ή τροποποίηση της οδηγίας πλαισίου, όπως γνωρίζετε, σας το λέω μάλλον, τώρα τελειώνουμε μια μελέτη αντικτύπου των διαφόρων δυνατήτων χρήσης των βιοαποβλήτων, το αναφέρει και το Green Paper, εξετάζουμε τα υπέρ και τα κατά, κάθε νομικού εργαλείου για να δούμε πώς θα πετύχουμε καλύτερα το στόχο μας. Δεν έχουμε διαμορφώσει λοιπόν άποψη. Ολοκληρώνουμε όπως σας είπα την μελέτη αντικτύπου. Θα κάνουμε ένα κατάλογο των υπέρ και των κατά για κάθε νομικό εργαλείο. Ευχαριστώ. Κύριε Τσίτσεστερ, θέλετε να πείτε κάτι? Να απαντήσω στο αίτημα για να υπάρξει χωριστή οδηγία. Χαίρο που ακούω ότι η Επιτροπή το σκέφτεται ακόμα. Είναι σημαντικό να το λάβει υπόψη, αλλά θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη και άλλες διαστάσεις. Ας προχωρήσουμε λίγο πιο προσεκτικά. Να σας πω τη δική μου εμπειρία στην πατρίδα μου στην νοτιοδυτική Αγγλία όπου γίνεται διαχωρισμός ε, αποβλήτων και έχουν προσπαθήσει, έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε διάφορες μορφές συλλογή των ε, ε, σκουπιδιών, δηλαδή τα βιοαποδομήσιμα τα μαζεύει ε, σκουπιδιάρικο κάθε δεκαπενθήμερο, άλλες ε, επικίνδυνα προϊόντα τα μαζεύει μια φορά την εβδομάδα. Δεν, έχουμε διάφορες ε, δυνατότητες. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα. Αν ξεκινήσουμε μια νομοθετική ρύθμιση όλων των ειδών βιολογικών αποβλήτων μπορεί να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσουμε. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε σε οικογενειακό επίπεδο, να κάνουν κομποστοποίηση ας πούμε, να χρησιμοποιούν ε, τα βιο απόβλητα με τρόπο που να επανέρχονται στο έδαφος και αν αντίθετα υιοθετήσουμε ένα καθεστώς ε, που καλύπτει όλα τα βιολογικά απόβλητα, νομίζω ότι υπερβαίνουμε την αναγκαία νομοθετική προσέγγιση. Πιστεύω ότι αφήνοντα την άκρη το κομμάτι εκείνο των αποβλήτων που δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να εξαφανίσουμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την πραγματική εκμετάλλευση των βιολογικών αποβλήτων. Αυτό είναι αναγκαίο. Τώρα αν χρειάζεται νομοθετικό κείμενο ή όχι δεν είμαι τόσο σίγουρο. Περιμένω την γνωμοδότηση τη συναδέλφου. Προσωπικά δεν είμαι αντίθετο, αλλά δεν καίγομαι κιόλα. Τώρα το χρονοδιάγραμμα πρόεδρε. 17 Μαρτίου τροπολογίες. Μέχρι τι 17 Μαρτίου. Όχι. Άλλαξε. Α. 25 Φεβρουαρίου. Αυτή τη βδομάδα. Το μεσημέρι βεβαίως. Η ψηφοφορία είναι το Μάρτιο. Ευχαριστώ, δεν ζητάει κανένα άλλο τον λόγο. Τελειώσαμε για σήμερα το πρωί. Τα λέμε το απογευματάκι. Γεια σας.